Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε. Μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης, η έκθεση Tech Talkers για τον εξυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της Ευρώπης. Τέσσερα λεπτά έχει ο εισηγητής. Με συγχωρείτε που καθυστέρησα κύριε Πρόεδρε, αλλά νόμιζα θα ξεκινούσαμε 10 λεπτά αργότερα. Θα παρουσιάσω την, την ομιλία μου ουγγαρέζικα. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για μια μεγάλη τιμή για μένα που μπορώ να σας μιλήσω για τον εξυγχρονισμό της σχολικής επέδευσης στην Ευρώπη καθότι είμαι εισηγητής επί του θέματος. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και τους συμβούλους, τους σκιώδης εισηγητές την Επιτροπή Γυναικών, τις αγαπητές συναδέλφους και την Επιτροπή την Περιφερειακή, την Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και ορισμένους οργανισμούς που με βοήθησαν πολύ. Ευχαριστώ για τη στενή συνεργασία διότι συνέβαλαν στο να μπορέσω να καταρτήσω την έκθεση αυτή και θεωρώ ότι το έργο του η συγητή είναι πάντοτε πολύ λεπτό και εγώ προέρχομαι από την Ανατολική Ευρώπη από μια χώρα η οποία πρόσφατα προσχώρησε ε, στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και όπου στο παρελθόν ε, στη Ρουμανία δεν θα μπορούσε να υπάρξει ένα πανεπιστημιακό σύστημα. Δεν υπήρχε η, καμία ανεξαρτησία, δεν γίνονται αποδεκτές ιδεολογίες και διαπιστώνω ότι γιατί τις χώρες ε, της Ανατολικής Ευρώπης ε, οι οποίες προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσφάτως είναι πολύ σημαντική, σημαντικός ο εξυγχρονισμός ε, του πανεπιστημιακού συστήματος διότι πρέπει να επιλύσει κανείς πολλά προβλήματα να καλύψει το κενό το οποίο υπήρχε με τη Δυτική Ευρώπη και να προσεγγίσουμε στο πανεπιστημιακό πανεπιστημιακό χώρο τα ε, πανεπιστήμια της Δυτικής Ευρώπης. Είχαμε πάρα πολλές τροπολογίες, κάπου 190, οι οποίες υπευλήθηκαν και οι οποίες αναφέρουν ότι κατόπιν της κρίσεως πρέπει να εξυγχρονίσουμε το πανεπιστημιακό μας σύστημα. Είναι μία επιταγή και γι' αυτό η έκθεσή μου αναφέρεται σε αυτόν τον εξυγχρονισμό και αναφέρουμε ποιες είναι οι προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να μπορέσουμε να λύσουμε τα υπόλοιπα προβλήματα δημοσιονομική έλλειψη πόρων, ποσοστό ανεργίας, δημογραφική κρίση που πλήττουν το, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί κανείς να προωθήσει τα θέματα αυτά και ε, το σύνολο αυτό των πανεπιστημίων παίζει μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στην έκθεση αυτή αναφέρεται ότι τα πανεπιστήμια θα πρέπει να συνεργαστούν με τους υπόλοιπους εταίρους τους, με ε, τους δήμους, με τους ε, πολίτες, με όλα τα, τις ομάδες συμφοερώντων σε όλους. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα ασχέτως της πολιτικής τους ή κοινωνικής τους προελεύσεως. Θα πρέπει να καταφερθούμε κατά των διακρίσεων και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει η πολυγλωσία και ότι θα μπορέσουν να υπάρχουν κοινωνικές κατά τρόπον ώστε οι εθνικές και γλωσσικές μειονότητες να μπορέσουν να διατηρηθούν, τα συμφέροντά τους να ε, ε, προσπιστούν και ε, θα τελειώσω την έκθεσή μου αναφερόμενος στην νεολαία διότι στις μετακομμουνιστικές χώρες βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό της ανεργίας των νέων και ελπίζουμε ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές μαζί με την έκθεση Berlinguer του Μαρτίου με την δική μου έκθεση και με άλλες εκθέσεις θα συμβάλλουν στην ε, εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής του 2020 και ότι θα μπορέσουν οι νέοι να βρουν δουλειά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ξεπεράσατε το χρόνο ομιλία σας κατά ένα λεπτό. Τώρα αρχίζει η διαδικασία του Catch the Eye. Έχουμε 12 εγγεγραμμένους ήδη στον κατάλογο των ομιλητών. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε τον χρόνο ομιλία σας για να μπορέσω να δώσω το λόγο σε όλους σας, μια και ήρθατε να συνεδριάσουμε τόσο αργά στην Ολομέλεια. Αλλά σας παρακαλώ να είσαστε συντομότατοι. Ευχαριστώ. Πρώτος ομιλητής λοιπόν, ο κύριος Βέρ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Τόκες για την εξαιρετική έκθεση διότι πρόκειται για μία εξαιρετική όπως είπα έκθεση και είναι μία νέα απόδειξη για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να βελτιώσουν ε, το πανεπιστημιακό σύστημα στην Ευρώπη. Ε, πάντοτε στην Ευρώπη υπήρχε ένα λίκνο της ε, προόδου των αξιών και του πολιτισμού και μπορούμε να μιλήσουμε για την τρίτη αποστολή της, ε, του σύμπαντος γι' αυτό και πρέπει να ανοίξουν τα πανεπιστήμια να υπάρχει καλύτερος διάλογος μεταξύ τους να υπάρχει μία δημοσίευση όλων των γνώσεων οι οποίες χρειάζονται κατά τρόπον ώστε ε, να βελτιωθούν και τα προγράμματα και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ εις ε, το όργανο το οποίο θα καταρτιστεί και θα πρέπει να είναι καλύτερο από ό,τι τα ισχύοντα. Παρακαλώ περιορίστε το χρόνο σας, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να παρέμβουν όλοι οι ομιλητές. Η επόμενη είναι η κυρία Τσίσκοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε σχέση με αυτή την έκθεση θα ήθελα να υπογραμμίσω την επιτυχία του προγράμματος Εράσμους που ε, βοηθάει την κινητικότητα των φοιτητών. Θα ήθελα ακόμη να τονίσω ότι αν πρόκειται να ανταγωνιστούμε με τις ασιατικές χώρες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πλήρως ε, το δυναμικό πολλών τεχνικών ε, επαγγελμάτων. Ακόμη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και το δυναμικό πολλών γυναικών που είναι δραστήριες στην έρευνα και την ανάπτυξη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος όταν επιλέγουμε ένα μάθημα πανεπιστημιακό να επιβάλλουμε διακρίσεις κατά των γυναικών. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, κάποια παραδοσιακοί ρόλοι για τα δύο φύλλα και κάποια στερεότυπα. Εντάξει, αλλά είμαι πεπισμένη ότι πρέπει να καταργήσουμε αυτά τα εμπόδια και αυτό θα είναι εφικτό μόνο με τη βάση ποσοστώσεων. Τα έλεγα λοιπόν ε, από την άλλη πλευρά είμαι κατά τέτοιων ποσοστώσεων και δεσμευτικών μέτρων. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Βασέσκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χρειαζόμαστε ανταγωνιστικά πανεπιστήμια στην Ευρώπη η προσφορά πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Υποστηρίζω την ιδέα συσχετισμού της ε, εκπαιδευτικής προσφοράς των πανεπιστημίων με τις ευκαιρίες απασχόλησης. Σύμφωνα με το άρθρο 27, ε, ε, ο αριθμός των φοιτητών στην Ρουμανία τετραπλασιάστηκε τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν μπορούν να βρουν δουλειά μετά που να ανταποκρίνεται στα προσόντα τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν προγράμματα για την πρώτη θέση εργασίας και για την ε, συνεχή κατάρτιση. Θα ήθελα ακόμη να αναφερθώ στο γεγονός ότι οι ενώσεις των φοιτητών δεν είναι ικανοποιημένοι με το Εράσμους. Η κριτική τους αφορά τις ελλείψεις, την τυπική εκπαίδευση, την έλλειψη διαδραστικής παιδείας.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

ε, περιλαμβάνει διάφορα σημαντικά θέματα αναφέρεται στην αυτονομία των πανεπιστημίων συρίζει το πρόγραμμα Έρασμος αναγνωρίζει τα διπλώματα και ε, επίσης ε, θέλει να εφαρμόσει την Επιτροπή Καλής Γειτονίας με τους γείτονές μας και δεν περιορίζεται στη στήριξη της οικονομίας. Υπάρχουν όμως και ανησυχητικά πράγματα όπως παραδείγματο χάρη η τυποποίηση του προγράμματος των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, υποχρέωση να, ε, να φοιτεί κανείς ένα εξάμεινο εκτός του πανεπιστημίου του. Η κυρία Ρούπερτ είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Πορτογαλία το σχέδιο της Μπολόνια και ο εξυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκάλεσε πολλές καταστροφές. Αντί να υπάρξει μια κινητικότητα των φοιτητών, προέκυψε μια ελίτ που δημιουργήθηκε στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Υπάρχουν φοιτητές που τελειώνουν το πανεπιστήμιο και που δεν καταφέρουν ε, να κερδίσουν τα προστοζήν. Ε, δεν καταφέρουν να πάρουν πτυχίο γιατί δεν έχουν καμία χρηματοδότηση. Εδώ μιλάτε για ένα πραγματικό αντικατοπτρισμό στην ουσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ευρωπαϊκή οικονομία μπορεί να αφήσει πίσω της την οικονομική αυτή κρίση αν εστιάσουμε την προσοχή μας στο εκπαιδευτικό σύστημα και ιδιαίτερα τη συνειδητοβάθμιση εκπαίδευση όπως προβλέπει το πρόγραμμα 2020. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να γίνει πιο ανταγωνιστική η οικονομία μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι όμως ε, επαρκές το να έχουμε πιο ικανά ε, πιο καλά πανεπιστήμια. Θα πρέπει να μπορούν ε, οι απόφοιτοι να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, γιατί στον τομέα αυτό είναι δύο φορές πιο υψηλή η ανεργία. Το πρόβλημα της ποιότητας είναι επίσης σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται ένας ενιαίος μηχανισμός, ο οποίος θα αξιολογεί τα ακαδημαϊκά πρότυπα σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσώπων στην Ευρώπη, γιατί αυτό οδηγεί σε μια μεγαλύτερη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, εισηγητή για την έκθεση αυτή που είναι πάρα πολύ σημαντική για τι επερχόμενε γενιές. Ευχαριστώ. Ο κύριος, η κυρία Σνεμιντέλοβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ε, ευχηθώ καλό βράδυ σε όλους το, τους παρισταμένους διότι κανείς ε, δεν, ε, δεν φέρει αντίρρηση σε μία βελτίωση των πανεπιστημίων χρειαζόμαστε καλά κατηρτισμένους φοιτητές και θα πρέπει να συμβάλλουμε και στο οι γυναίκες να έχουν καλύτερη πανεπιστημία πανεπιστημιακή παιδεία, χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες στα πανεπιστήμια για να μπορέσουν να έχουν καλύτερες ευκαιρίες και να μπορέσουν να συμβάλλουν περισσότερο στη ζωή της κοινωνίας τους. Θα πρέπει να τη στηρίξουμε και να στηρίξουμε και τη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων. Μια άλλη σκέψη που είναι πολύ σημαντική για μένα είναι ότι αναφέρουμε τις ε, ε, χορηγήσεις και τα δάνεια και θα πρέπει να σκεφτούμε και τους κοινωνικά υστερούντες. Ο κύριος Κέλλη. Θα μπορούσα να μιλήσω όλο το βράδυ ε, ε, με πρώην εκπαιδευτικό, αλλά δεν υπάρχει χρόνο. Είναι μια από τι καλύτερε προτάσει που είχαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγχαίρω λοιπόν τον εισηγητή και την Κομισιόν. Είναι πρόκληση για τα τριτοβάθμια ιδρύματα για να ανταποκριθούν στο στόχο του 2020 40% θέλουμε των παιδιών, των νέων να, πάνε στην, να αποφυτίσουν από την βάθμια. Είναι πρόκληση αυτό και βεβαίω στη σχέση στη συνέχεια πρέπει να διασυνδέσουμε τα πτυχία με την αγορά εργασία αν πρόκειται να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ε, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα τώρα. Βεβαίως, η ισότητα των φύλων είναι απαραίτητα απαραίτητη και είναι γελίο για ιδρύματα που θεωρούν ε, ότι είναι τα καλύτερα στον κόσμο να μην σέβονται αυτή την ισότητα. Τέλος θα ήθελα να κάνω το εξή σχόλιο. Να μην μιλάμε πια για καθηγητές και λέκτορες. Είναι δάσκαλοι. Δάσκαλοι διδάσκουν τα παιδιά. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Παπανικολό. Να συγχαρώ και εγώ τον εισηγητή για την εξαίρετη δουλειά του διαβάζοντας την έκθεσή του αλλά και την στρατηγική μας για την ευρώπη για το 2020 όλοι συμφωνούμε ότι είναι ανάγκη να επενδύσουμε στην παιδεία αλλά και να αυξήσουμε το ποσοστό των αποφύτων των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Απ' την άλλη όμως βλέπουμε την ίδια περίοδο και πραγματικές μειώσεις έως και 10% στις κρατικές δαπάνες πολλών κρατών μελών για τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδίων μάλιστα αυτών που βρίσκονται ε, υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης ε, οι χώρε του Νότου σοβαρέ αντιφάσει λοιπόν ανάμεσα στου στόχου στι διακηρύξει και στι πράξει. και επειδή η παιδεία και ο εξυγχρονισμό τη αυτά που συζητάμε σήμερα δηλαδή δεν είναι ζήτημα διαπιστώσεων αλλά πρακτικών αποτελεσμάτων επειδή η επένδυση στο τρίγωνο τη γνώση αποτελεί προτεραιότητα για την ανάταξη των εθνικών οικονομιών θα ήθελα να ρωτήσω και την επιτροπή που βρίσκεται σήμερα εδώ αν σκέφτεται να προτείνει στα κράτη μέλη να εξαιρέσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση από τι γενικέ περικοπέ στι δημόσιε δαπάνε ή αν θα προτείνει αντισταθμιστικά μέτρα διότι ακούγεται στου πολίτε παράλογο και δικαίω να μιλάμε από τη μία για εξυγχρονισμό ενώ παράλληλα να περικόπτονται μαζικά πόροι από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ διότι άκουσα το, είδα το όνομα του κυρίου Τέκες που ανέλαβε αυτή την ε, εκθεσή και είναι ένας ε, ε, επίσκοπος ε, ο οποίος φρόντισε ε, να περιλαμβάνεται στην έκθεσή του οι αρχές του χριστιανισμού και η εκπροσώπηση των ε, συμφερόντων των μειονοτήτων στην Ευρώπη. Αλλά από τα 77 σημεία μόνο ένα αναφέρεται εις τα πανεπιστήμια για τις μειονότητες και μόνο ένα στην ισότητα των και θεωρώ ότι αυτό είναι άνισο διότι δεν ε, μπορούν όλα να λειτουργήσουν όπως το Βέλγιο που υπάρχουν ε, δίγλωσσα σχολεία στη Ρουμανία ε, δεν έχουμε ευχέρεια για εκπαίδευση των Ουγγροφόνων και γι' αυτό δεν θα στηρίξω την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, χρειάζεται μία δυναμική ανάπτυξη των πανεπιστημίων για να μπορεί να προωθηθεί η κοινωνία και δεν είναι μόνο θέμα γροήτρου, αλλά και προϋπόθεση για να βρει κανείς μία θέση εργασίας. Παρόλα αυτά όμως βλέπουμε ότι η δεν ε, ε, ανταποκρίνονται οι προσφορές στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο στο μέλλον κατά τρόπον ώστε τα πανεπιστήμια να προσαρμοστούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας για να μπορέσουμε να ε, δούμε μία ισορροπημένη ανάπτυξη και θα πρέπει να προωθηθούν μόνο τα ιδρύματα όπου οι απόφοιτοι μπορούν στη συνέχεια να βρουν θέση ή στην κοινωνία και γι' αυτό θα χρειαστούν καλύτερα κριτήρια επιλογής. Τελευταίος ομιλητής ο κύριος Τζόκα. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για αυτή την έκθεση. Είναι αλήθεια ότι καθημερινά έχουμε να αντιμετωπίσουμε πήγοντα ζητήματα, αλλά σήμερα μιλάμε για οριζόντια θέματα ε, και μπορούμε να κοιτάξουμε τα αποτελέσματα για τις μελλοντικές γενιές. Η μοντέρνα Ευρώπη έχει τις ρίζες της στην εκπαίδευση των νέων. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να μεταρρυθμίσουμε ολόκληρο το σύστημα. Τα πανεπιστήμια παίζουν ρόλο κλειδί. Τα πανεπιστήμια όμως δυστυχώς δεν είναι ανταγωνιστικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι το Youth in Action σαν πρόγραμμα θα πρέπει να θεωρηθεί σαν σημαντικό εργαλείο. Χρειαζόμαστε καινοτομία σε σχέση με την έρευνα και πάντοτε σε συνδυασμό με την αγορά εργασίας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις μελλοντικές διαρθρωτικές πολιτικές να εξυγχρονίσουν τα πανεπιστήμια. Πρόεδρος. Και τώρα δίνω το λόγο στον Επίτροπο. Καλ... Καλωσορίζω εκ μέρου της Κομισιόν την έκθεση του κ. Τάκο. Καλωσορίζω την φωνή του Ευρωκοινοβουλίου πάνω σε αυτό το θέμα. Χαίρομαι που δίνεται προτεραιότητα και είναι επίκαιρο το ζήτημα διότι αφενός κανείς δεν αναγνωρίζει ότι η οικονομία με βάση τη γνώση είναι το μέλλον της Ευρώπης και από την άλλη πλευρά η λιτότητα σημαίνει περικοπές σημαντικές στους εκπαιδευτικούς προϋπολογισμούς. Θέλω να απαντήσω στον κύριο Παπα-Νικολάου. Επανειλημμένως τονίζουμε ότι ακόμη και σε περίοδο λιτότητας η κατάρτιση παιδεία πρέπει να τυχαίνει ιδιαίτερα θετικής μεταχείρισης στον προϋπολογισμό. Αλλιώς υπονομεύουμε το μέλλον της Ευρώπης. Επίσης γνωρίζουμε το παράδοξο της σημερινή Ευρώπης, δηλαδή ότι έχουμε σχετικά ε, εργατικό δυναμικό με υψηλά προσόντα στην Ήπειρό μας, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε διαρθρωτική ανεργία, ε, ιδίως όταν έχουμε να κάνουμε με αυτό που αποκαλούμε ήδη τη χαμένη γενιά. Άρα, η διασύνδεση μεταξύ παιδείας και αγοράς εργασίας είναι περίπλοκη και χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις ε, για να πετύχουμε ολοκληρωμένο ανταγωνισμό τα προσόντα, τα σημαντικά, θα, είναι, θα παίξουν τον σπουδαιότερο ρόλο στο μέλλον, αλλά πρέπει να συμμετέχει και ο επιχειρηματικός κόσμος και οι άλλοι μας εταίροι, ώστε οι απόφοιτοι της βάθμιας να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά και χρειαζόμαστε και επαγγελματικά προσόντα πολύ συγκεκριμένα για να αποφύγουμε την ανεργία. Στην έκθεση του κυρίου Τέκες η ατζέντα που που προτάθηκε από την Κομισιόν το Σεπτέμβριο του 2011 υποστηρίζεται για την καινοτομία και την τεχνολογία. Έχουμε πολυδιάστατη προσέγγιση για τη βαθμολόγηση των πανεπιστημίων. Έχουμε ακόμη την πρόταση για ορισμένες συμμαχίες τρόπων την άμεταξη ε, Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας και δεν πρέπει να υπονομεύσουμε τους προϋπολογισμούς των προγραμμάτων των μελλοντικών όπως του Erasmus for All, του Marie Curie κτλ. Και το Erasmus για το Erasmus προτείνεται από την Κομισιόν μια εγγύηση για δάνειο που να βοηθάει τους φοιτητές εκτός από την επιδότηση που δίνεται. Ε, στον φοιτητή. Και βεβαίως για το μέλλον δεν θέλουμε μόνο μαζικά να ενισχύσουμε την παιδεία, αλλά θέλουμε να δημιουργήσουμε και εταιρικέ σχέσεις μεταξύ ιδρυμάτων. Σας ευχαριστώ κύριε Τόκερς και πάλι για την θετική προσέγγισή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελείωσε η συζήτησή μας και η ψηφοφορία προβλέπεται για αύριο στις 12. Το τελευταίο σημείο της